everyone. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, μάμα. Παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας. Ο κύριος Μπουσόη ξέχασε την κάρτα του, οπότε θα μας επισημαίνει κάθε φορά την ψήφα του μέχρι το έρθει η κάρτα ψηφοφορίας. Έχετε υπόλοιποι της ε, ηλεκτρονικές κάρτες. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε το πρώτο θέμα που είναι σχέδιο ψηφίσματος για την ε, ε, έγκριση κάποιων χρήσεων για το διχρωμικό νάτριο με βάση τον κανονισμό 907 του 2006. Μία και μόνο ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ο κύριος Μπουσόη αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η αντίρρηση. Δεύτερο θέμα. Σχέδιο έκθεση με, με βάση μια πρόταση κανονισμού που προβλέπει τη θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και την κλιματική δράση, το πρόγραμμα LIFE και την κατάργηση ενός κανονισμού του 2013. Ξεκινάμε με κάποιες ταυτόσιμες τροπολογίες 162-163 και Ρεγί 22. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, με μπέρδεψαν. Οι σοσιαλιστές είναι διχασμένοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 164. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Καταπίπτει, συγγνώμη. Καταπίπτει. Το ίδιο και η 23 της Ρέγγι. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 27 υπέρ και 42 μαζί. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτονται. 169. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 6. Συμβαστική τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 198 και 199 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 201, Ρέτζι 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. 202. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ? Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως πρώτα για την τροπολογία 202. Άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Μπουσό, έχετε πια την κάρτα σας. Μάλιστα. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται η 202. Συμβαστική τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 11. 36 της Ρέντζη. Ποιος είναι υπέρ. 36 της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κατά αποχές απορρίπτεται. 244. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 244. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 245 και 247 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 246. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται 37 και 21 της Ρέτζη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 249 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18. ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ. Τροπολογία 264 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 268 καταπίπτει. 271. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 275 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 277 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η πράσινη ήταν υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 18 και στην τροπολογία 285 και άγκρι 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 300. Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως πρώτα. Μα μόνο το ΕΛΚ και το ECR ήταν υπέρ. Αλλά αν, να το ελέγξουμε αν προτιμάτε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 285 και άγκρι 26. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Λυπάμαι κυρία η δική σας ήταν η τροπολογία, εγώ την υπερψήφισα. Αλλά δεν τελεσφόρησε. 300, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 301 και άγκρι 30, ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για αυτές. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ίδια διαφορά, μία ψήφος διαφορά. Απορρίπτεται όμως, απορρίπτονται. 302, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 36, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος και εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά αυτή τη φορά. Ενδιαφέρον. Ρέγγι 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 304. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Αλλάζουν οι πλειοψηφίες. Ανάλογα με την τροπολογία, άλλες περάνε και άλλες όχι με μία ψήφο διαφορά. Πάμε στη σελίδα 21. «326. Ποιος είναι υπέρ» Κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε κακού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Όντως απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. 13 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ποιος είναι υπέρ της 13. Α, ήταν βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η ομάδα σας, γιατί πέφτουν τροπολογίες υπέρναμε μια ψηφοδιαφορά. Ποιος είναι υπέρ της budget 13, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 21, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 51 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 333, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 339 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 340. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 341 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 342 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 343 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 344 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 345 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 352 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 352 άρχεται η ψηφοφορία. Το ECR ε, τάχθηκε υπέρ, κάτι που με μπέρδεψε και τώρα βλέπω ότι καταψηφίζεται. Α, εσείς ψηφίσατε υπέρ. Α, μάλιστα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. εγκρίνεται. 356 υπέρ. Κατά. αποχέ, απορρίπτεται. 357 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 357 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται. 358, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 68 θα έλεγα ότι εγκρίνεται, αλλά δεν ε, σηκώσετε εμφανώς τα χέρια. Τέλος, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 80. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123. Υπέρ, κατά, αποχές, Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 15 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 70 ή μάλλον καταπίπτει 77. 139. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 17 ποιος είναι υπέρ. Η γραμματεία μου είπε ότι από τη στιγμή που η 203 απορρίφθηκε δεν ψηφίζουμε είναι 151. Ποιος είναι υπέρ της 17 κατά αποχές εγκρίνεται. 150, ή μάλλον και αυτή καταπίπτει, 153, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 161 άρχεται η ψηφοφορία ίσως εγκριθεί με δυο ψήφους διαφορά. Σας τα είπα. Πραγματικά εγκρίθηκε με δύο ψήφου διαφορά. 63. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία. Ή ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης σε ψηφοφορία για την πρόταση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας και την κατάργηση του ε, κανονισμού. Ξεκινάμε με την τροπολογία 117. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά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 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ. Είναι ψηφοφορία unblock. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134, πάλι unblock, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135, block, C, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 136, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 137, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 143, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 146, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 12 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Οι πράσινοι απέχουν πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 154. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά δεν σηκώνω τα χέρια. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάλι με μία ψήφο παραπάνω. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κύριε Ντάνις, πώς ψηφίσετε. Υπέρ. Α. Ψηφοφορία Κατά τμήματα θα ελέγξουμε 159. Ή δεν είναι κατά τμήματα. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Παλούτσι. Πέρας. Εγκρίνατε. Πάλι με μία ψήφο παραπάνω. 160. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 163. Καταπίπτει 163. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 και 164. Υπέρ. Κατά. Φιλελεύθεροι, δεν μπορείτε να είστε ταυτόχρονα υπέρ και κατά. Πάλι από την αρχή. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 και 168 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέρας πληροφορίας. Μάλιστα, το ΕΛΚ λοιπόν είναι διχασμένο βλέπω. Και πάλι εγκρίνεται με μία ψήφο παραπάνω. Τουλάχιστον τρεις καταψήφισαν. Όμως εγκρίθηκε. 178 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο στην 183. Πέρας. Εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Τι περίεργο συνδυασμό είναι αυτός. Τι κάνουμε τώρα. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. την 19. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάλι με μία ψήφο. Σήμερα είναι δύσκολες οι ψηφοφορίες. 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187. Υπέρ κατά αποχές απέχουν οι πράσινοι. Έλεγχος λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά Δεν βλέπω το έλγη, να σας πω την αλήθεια. Ξανά, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Μένει ένας να ψηφίσει, τώρα ψήφισαν όλοι, εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 195. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 196. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το υπέρ. Ναι. Ωραία εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 201 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 202 υπέρ κατά φιλελεύθερη είναι υπέρ εγκρίνεται 203 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σε block D. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 μπλοκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 218 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπλοκ 219 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές φιλελεύθεροι, ίσως είστε διχασμένοι. Να το κοιτάξουμε. 17, άρχεται ψηφοφορία. Έτσι φαίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 70. Ψηφίσατε όλοι, γιατί Είμαστε πολλοί. Α, πέρας. Εγκρίνεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. ECR. Είστε υπέρ. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάλι με τον ίδιο αριθμό ψήφων. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Δεν μας δείξατε κάτι. Πέρας. Εγκρίνατε. Δεν έχουμε πολλές ψηφοφορίε. οπότε αν μου δείξετε τι θέλετε, δεν χρειάζεται να ελέγχουμε κιόλας. 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 76 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 81 άρχη ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο τη τροπολογία. 4. Άρχεται η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 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 108 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε ένα συντομότερο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πιέκα. Σχέδιο γνωμοδότησης για μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνική νοημοσύνη και τη ρομποτική. Τροπολογία 28 εγκρίνεται, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται, αλλά για να είμαστε σίγουροι, επειδή είναι συμβιβαστική, να ελέγξουμε. είναι συμβιβαστική. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37. Ποιος είναι υπέρ του 37. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές υπέρ. εγκρίνεται. 52. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Ψηφίσουμε το πρώτο μέρος ψήφι υπέρ του πρώτου μέρους κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές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 άρχια η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έγκριση τροπολογιών για τις για τους δείκτες αναφοράς ε, για τη χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Ελέγχουμε την τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε το 25. Αρχή της ψηφοφορίας.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42, 43 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 44, 45 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Για να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες του κυρίου, ε, την κυρία Πιεντικάνεν, συμπεριλαμβανομένης και της 58.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 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Μετά 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21, 22, 23 ψηφίζουμε όλες μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Now we are voting again. Ξαναψηφίζουμε μια έκθεση και τις τροπολογίες ό,τι αφορά την θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Εδώ είναι πολύ δραστήριος ο κύριος Φλάναγκαν. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε συλλήβδια μερικές τροπολογίες Φλάναγκαν. 34. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 40 άρχεται η ψηφοφορία Απορρι... Ε, ολοκληρώνεται και απορρίπτεται 41 και 42 Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 με 61 γίνονται όλες μαζί. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτονται. 62 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 1 με 3, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτονται. 4 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 με 16. Όχι μαζί. 12 με 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά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 κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ 31 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Και τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και η τελευταία μας ψηφοφορία τώρα. Ψηφίζουμε πάλι και μια έκθεση με τη μορφή τροπολογιών που αφορούν την, σήμανση, την επισήμανση των επισώτρων με σεβασμό της αποτελεσματικότητας των καυσίμων και άλλων συναφών παραμέτρων και κατάργηση κανονισμού του 2009. 28. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 31 τέλος εγκρίνεται 32 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά. Η πράσινη είναι υπέρ ή κατά. Εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μαζί με τη 37 ήταν αυτή. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές δεν καταλαβαίνω το αποτέλεσμα. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 39. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τελικά. Τροπολογία 40. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές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 Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες το απόγευμα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρον απόγευμα με τον δόκτωρα Τάντρο, τον Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας θα έχουμε και την εκδήλωση της υπογραφής που θα μας παρουσιάσει το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Υγεία. Θα έχουμε και μια πανηγυρική εκδήλωση με την υπογραφή. Πραγματικά, ελάτε. Αν δεν έρθετε για τον δόκτωρ Γκέντρος, για ποιον θα έρθετε πια. Στις 5 θα έρθει ο καλεσμένος μας, αλλά θα προηγηθούν κάποιες ψηφοφορίες στην αρχή της συνεδρίασης. Καλή σας όρεξη.